Ε, εξετάσουμε αυτή την έκθεση και θα δώσουμε απαντήσεις και στους εμπλεκόμενους φορείς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπη, σας ευχαριστώ συνάδελφοι που μείνατε τόσο αργά. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η συζήτηση έχει λήξει και η ψηφοφορία θα λάβει η χώρα την Τετάρτη. Η επόμενη συνεδρίαση θα, γίνει, θα αρχίσει αύριο στις 9. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευτεί στο διαδικτυακό μας τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.